Dear colleagues, please be seated so that we can... Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Thank you very much. So let me open... Σας ευχαριστώ και να ξεκινήσουμε λοιπόν την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Οικών και ΕΜΠΛ, Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και Απασχόλησης, ένα σημείο μόνο στην ημερήσια διάταξη και να ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη και την έγκριση αυτή. Δεν βλέπω σχόλια και ενστάσει. Ε, να περάσουμε λοιπόν στο πρώτο σημείο. Οικονομικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων για την ετήσια έρευνα ανάπτυξη και για τον στην αναφορά του μηχανισμού ειδοποίηση, με τον Βάλτε Δομπρόσκη, και Αντιπρόεδρο και τον κύριο Πιχέρη Μοσκοβισή, Επίτροπο. Εγώ αντικαθιστώ τον κύριο Κουτιέρη, τον πρόεδρο τη Επιτροπή μα ο οποίο θα καταφτάσει λίγο αργότερα. Καταρχάς, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο, τον και τον Επίτροπο Μοσκοβισή για τον οικονομικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων για την ετήσια έκθεση ανάπτυξη και το μηχανισμό επαγρύπνηση. Να σα υπενθυμίσω ότι η, η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί τμήμα του, της διαδικασίας που ορίζεται στον κανονισμό Six Pack και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε την πρόταση για το Six Pack στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου και ο οικονομικός αυτός διάλογος και οι εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές των εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων ίδιας πρωτοβουλία και της κοινή ε, έκθεση από πλευρά της Επιτροπής Απασχόλησης ανέκριναν πριν από την Σύνοδο της Άνοιξης την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο προκειμένου να υπάρξει λογοδοσία στην, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των, ε, της έκθεσης αυτής και έτσι η ετήσια έκθεση 2018 ε, δίνει το ένα αυτό για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ορίζοντα τόσε ευρείε οικονομικέ προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το επόμενο έτο. Και όπω έγινε και πέρσι, συνοδεύεται από συστάσει για την σύσταση του Συμβουλίου για την οικονομική πολιτική της, του χώρου ευρώ για να ενσωματωθεί καλύτερα ο χώρος του ευρώ και τα εθνικά επίπεδα του ευρωπαϊκού εξαμένου. Και έτσι λοιπόν στη σειρά θα είναι όσο ακολουθεί. Ως εξής τι εισαγωγικά σχόλια από πλευρά τη Επιτροπή ε, θα τα μοιραστούν ο Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκη και ο Επιτροπό Μοσκοβίση. 15 λεπτά σα παρακαλώ, μην τα υπερβείτε. Και μετά θα έχουμε γύρω ερωτοπαντήσεων από τα μέλη τη Επιτροπή Οικονομικών και Απασχόληση. Ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στον κύριο Ντομπρόφσκη. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ. Όπως Ήδη μας ε, είπατε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πακέτο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το προηγούμενη εβδομάδα και αυτό σηματοποτεί την έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2018 και έτσι περιλαμβάνεται η έρευνα αιτήσει ανάπτυξη που θέτει οικονομικές και πολιτικές και κοινωνικέ προτεραιότητε για το επόμενο έτη και τον μηχανισμό επαραγρύπνηση που επισημαίνει τους κινδύνους και τις ανισορροπίες που υπάρχουν στο κράτη-μέλη. Και έτσι έχουμε και την κοινή έκθεση από την Επιτροπή Επασχόλησης που συγκρίνει τις απαντήσεις και τις ανταποκρίσεις από πλευράς των ανακράτων μελών και τις συστάσεις για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, σύσταση για την περιοχή τη ζώνη ευρώ σε ό,τι αφορά τη διατύπωση εθνικών πολιτικών από πλευρά των εθνικών κρατών μέλων και 18 γνωμοδοτήσεις για τα μέλη της Ευρωζώνης σε ό,τι αφορά και τη σχετική ανακοίνωση. Το πακέτο μας λοιπόν έχει να καταδείξει την υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη της τελευταίας δεκαετίας. Όλα τα κράτη-μέλη αναπτύσσονται. Η απασχόληση έχει φτάσει σε ύψος ρεκόρ. Η ενεργία δε είναι σχεδόν ωστόσο χαμηλή όσο και πριν από την ε, κρίση. Οι επενδύσεις ε, ανακάμπτουν και τα δημοσιονομικά επίσης. Αυτό καταδεικνύει η στρατηγική μας η οποία βασίζεται σε τρεις βασικές ε, προτεραιότητες ε, επενδύσεις, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική δουλεύουν και επικεντρωνόμαστε λοιπόν στις προτεραιότητες αυτές και θα πρέπει να μείνουμε στον δρόμο αυτό γιατί εξακολουθούμε να έχουμε τις σημαντικές προκλήσεις η οριμότητα των αντιδράσεων διαφέρει από χώρα σε χώρα. Σε κάποιες χώρες έχουμε ακόμα υψηλή ενεργεία, τουλάχιστον για τους νέους και ε, μεγάλες ανισότητες και θύλακες προβληματικές, προβληματικούς στο τραπεζικό σύστημα. Η ανάκαμψη αποτελεί μια ευκαιρία να επιλύσουμε αυτά τα εκκρεμή ακόμα ζητήματα και τώρα λοιπόν θα χρειαστεί σε αυτού του καλούς καιρούς να οικοδομήσουμε μια στεναρή οικονομία, λιγότερο α, πιο αντακτική στους οικονομικούς κρατασμούς. Και θα πρέπει επίσης να υπάρξει και σύγκληση, θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη των οικονομιών, οι λιγότερο διμερείς θα πρέπει να αναπτυχθούν πιο γρήγορα και η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι συμπεριληπτική, να περιλαμβάνει όλους. Θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, με την αρχή τη ε, ισότητα και τη δικαιοσύνη, Σε ό,τι αφορά την αύξηση τη παραγωγικότητα, μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να πετύχουμε υψηλού όρου διαβίωση και ευημερία. Και προ την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να επενδύσουμε όχι μόνο σε υποδομέ, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό, στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Και επίση συστήνουμε στα κράτη-μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην παραγωγικότητα και στην αποδοτικότητα στι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει. Χρειάζεται μια καλή ε, αγορά εργασίας θα πρέπει να δίδονται οι σωστές ικανότητες και δεξιότητες στα άτομα και για τις ερχόμενες δεκαετίες εν ώψη και της, του διδάσκοντα πληθυσμού. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές για τα κρατημέλη που βρίσκονται σε διαδικασία διόρθωσης των μακροοικονομικών ανισοτήτων και ο μηχανισμός καταδεικνύει ότι τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα έχουν επιληθεί στα πιο πολλά κράτη-μέλη του 2016. Εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα φυσικά ανησυχία γιατί υπάρχουν ακόμα ζητήματα που καθιστούν ευάλωτα τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις χρειάζεται πολιτικό κεφάλαιο και θα πρέπει να δούμε ποια είναι το κόστος αλλαγής αυτών σε ό,τι αφορά την εμπειρογνωμοσύνη για την ε, εφαρμογή όλων αυτών των ε, διευθυντικών μεταρρυθμίσεων. Υπάρχει ένα πρόγραμμα όμως υποστήριξης των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δίδεται ακριβώς κάθε οδήγηση και στοχευμένη αρρωγή στα κράτη-μέλη εφόσον το ζητήσουν για να εφαρμόσουν αυτές τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις. Οι υπηρεσίε μα επίση υποστηρίζουν ήδη 15 κρατημέλη για 150 και πλέον τέτοια προγράμματα μεταρρύθμιση και στο νέο κύκλο έχουμε λάβει 144 αιτήματα από πάνω από 20 κρατημέλη. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από τη δημοσιονομική ικανότητα για το επόμενο έτος. Η τρίτη προτεραιότητα τη έρευνα τη ανάπτυξη είναι τα υπεύθυνα δημοσιονομικά, η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική βρίσκονται σε, σε διαφορετικέ φάσει του οικονομικού κύκλου τα κρατη και θα πρέπει να υπάρξει η σωστή ισορροπία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξη μεν τη ανάπτυξη και σωστά και βιώσιμα δημοσιονομικά η μείωση τη υψηλή χρέωση και ε, η δημοσιονομική πειθαρχία κάλυψη των κενών σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά και η καλύτερη στόχευση των ε, πόρων. Και επίσης ε, επισημάνετε αγαπητοί πρεβουλευτές τα θέματα τα κοινωνικά και τα θέματα της εργασίας. Ε, έχουμε και τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που παρουσιάστηκε και πριν από δύο εβδομάδες στο Κέντεμπορκ. Θα ήθελα να επενέσω το έργο του Κοινοβουλίου και της εισηγητρίας του κυρίου Ροντρίκες, για την, ε, της για την υποστήριξη προς τον πυλώνα αυτό. Προτείνεται λοιπόν να διορθωθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τα θέματα αυτά κοινωνικά και ένα νέο κοινωνικό scoreboard. Η απόδοση των κρατών μελών ε, αξιολογίζεται βάσει 14 δεκτών και προσμετράτε για παράδειγμα οι μεταρρυθμίσεις κοινωνικής πολιτικής βάσει των ε, στόχων που έχει θέσει και ο πυλώνας. Να κοιτάξουμε τώρα την Ευρωζώνη και τη σύσταση για την Ευρωζώνη. Επικεντρωνόμαστε σε βασικά θέματα για την καλή ε, λειτουργία της Ευρωζώνης, ε, αλλαγές προτείνονται για να υπάρξει σωστή και συμπεριληπτική ανάπτυξη και ανθεκτικότητα, ανθεκτικότητα και σύγκληση. Και Επίσης, προκειμένου να υπάρχει μια ουδέτερη δημοσιονομική στάση σε σχέση και με τα εθνικά τέτοιες εθνικές επιτροπές για την οικονομική ανάπτυξη και την εξέλιξη των δημοσιονομικών για, την, ε, για τα μέλη της Ευρωζώνης. Είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε προς μια EMU, μια οικονομική και νομισματική ένωση πλήρη αλλά όχι μόνο για αυτά τα κράτη-μέλη. Αυτό περιλαμβάνει και ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση και τη Ένωση κελφαλαγορών Αγορών. Και τους επόμενου μήνε θα καταθέσουμε μια πρόταση για να προωθήσουμε τα στοιχεία αυτή και θέλουμε να υπάρξουν διακυβερνητικέ ε, συμφωνίες στα πλαίσια του κοινωτικού πλαίσιου για, τον, για τη συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και το ESM θα πρέπει να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό προκειμένου να αντιμετωπίζουμε την κρίση με, καλύτερη, με καλύτερο τρόπο. Και επίσης περιλαμβάνονται ιδέες για ένα ευρωπαϊκό, ε, για μια ειδική, ειδικό κεφάλαιο στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό για την Ευρωζώνη σε ό,τι αφορά την αρρωγή των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων, τις ε, διαρθρωτικές αλλαγές αυτές, ε, ένα μηχανισμό σύγκλησης στον τομέα της Ευρωζώνης και ε, μια λειτουργία δημοσιονομικής σταθεροποίησης με, που προετοιμάσαμε και παρουσιάσαμε και τον Μάιο. και προστασία, αυτό περιλαμβάνει και η προστασία των ε, επενδύσεων. Γιατί σε περιπτώσει και περίοδου κρίση οι επενδύσει είναι αυτέ που πλήττονται πρώτε. Ε, να θυμόμαστε ωστόσο ότι η ενίσχυση του οικοδομήματο EMU δεν ε, μειώνει την ανάγκη δημοσιονομική πειθαρχία σε εθνικό επίπεδο σύγκληση, αλλά στο ιστορικό των κρατών μελών. Και εδώ λοιπόν είναι η ιδιαίτερη σημασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκη. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Επιτροπό Μοσκοβισή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με χαρά συμμετέχω σήμερα μαζί με τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκη σε αυτή τη νέα έκδοση του οικονομικού διαλόγου. η διαδικασία είναι σημαντική για τη διαφάνεια και το δημοκρατικό χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι προτάσεις πακέτο μας λαμβάνουν υπόψη στις συζητήσεις τις οποίες είχαμε μαζί σας με το Συμβούλιο, τα άλλα όργανα, τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τους κοινωνικούς εταίρους. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό το πακέτο είναι και το δικό σας πακέτο. Και φέτος έχει μια διαφορετική διάσταση για δύο λόγους. Πρώτον, αντικατοπτρίζει την διακήρυξη για τα ευρωπαϊκά θεμέλια των κοινωνικών δικαιωμάτων της συνάντησης κορυφής του Χέτεμπορχ το είπε ο Βάλτης. Απ' την άλλη έρχεται λίγες μέρες πριν από την παρουσίαση του πακέτου για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Να επανέλθω λοιπόν σε αυτό το πακέτο του φθινοπόρου του 18. Προτεραιότητα σήμερα είναι η ανάπτυξη, η οποία χαρακτηρίζει όλες τις χώρες μέρη, να είναι διαρκής και βιώσιμη και να ωφελεί όλους, όχι μόνο λοιπόν ανάπτυξη, αλλά μια ανάπτυξη μοιρασμένη, μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμό. Και το πακέτο μας δίνει τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή. Παρουσιάσαμε την προηγούμενη Τετάρτη την έκθεση για το μηχανισμό εγκαίρης προειδοποίησης η έκθεση αυτή είναι η εκκίνηση του ετήσιου κύκλου της διαδικασίας σχετικά με τις ανισότητες της μακροοικονομικές. Οι οικονομικές συνθήκες βελτιώνονται και αυτό βοηθά στην διόρθωση των ανισοτήτων που υπάρχουν σήμερα. Ε, πάντα ο αριθμός των χωρών για τους οποίους απαιτείται να υπάρξει ε, ένα σε βάθος αν θέλετε έλεγχος είναι απαραίτητο να φτάνει τις 12 και ε, θα δούμε, έχουμε ένα λιγότερο από ό,τι πέρυσι, η Φιλανδία δεν εντάσσεται στη διαδικασία αυτών των ανισορροπιών των δημοσιονομικών. Έχουμε λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας και το υψηλό επίπεδο χρέους ορισμένων χωρών. Είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επίσης υπάρχουν τα κόκκινα δάνεια που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα και επίσης ε, και η μείωση του εξωτερικού χρέους είναι κάτι το οποίο απαιτεί αρκετό χρόνο. Προτείνουμε λοιπόν 12 χώρες να ελεγχθούν ιδιαίτερα το 18 είναι οι ίδιες που ελέγξαμε την προηγούμενο κύκλο, Γερμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, κάτω χώρες, Πορτογαλία, Σλοβενία και Σουηδία. Για τις υπόλοιπες χώρες ε, δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται μια μελέτη σε βάθος, Υπάρχουν ε, στις εκθέσεις μας ορισμένα προβλήματα όπως ε, η απότομη άνοδος ε, της τιμής των ακινήτων και το κόστος του εργατικού δυναμικού. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες από πλευράς των χωρών οι οποίες έχουν ένα σημαντικό πλεόνασμα του ισοζυγίου πληρωμών για να επιτρέψουμε να γίνει αυτή η ρύθμιση στο σύνολο της ζώνης ευρώ. Απευθύνουμε λοιπόν για μια ακόμη φορά έκκληση στις χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν τα σημαντικότατα πλεονάσματά τους για να τονώσουν την εσωτερική ζήτηση και τις επενδύσεις. Είναι προς το δικό του συμφέρον και προς το συμφέρον του συνόλου της ζώνης ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει αυτές τις μελέτες στα πλαίσια των εκθέσεων αναχώρα το Φεβρουάριο του 2018. Να έρθω τώρα λίγο στη σύσταση τη σχετική με την οικονομική πολιτική της ζώνης ευρώ στο σύνολό της. Για πρώτη φορά φέτος οι συστάσεις μας που ζητούν από τα κράτη-μέλη να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους στα πλαίσια της καταπολέμησης των ευνοϊκών επιθετικών φορολογικών συμφωνιών. Υπεύθυνο Επίτροπος γι' αυτά είμαι εγώ και χαίρομαι για την πρωτοβουλία αυτή και ξέρω ότι και εσείς μας στηρίζετε στον τομέα των φυρολογικών πολλοί από εσάς συμμετέχετε εναργά στις εργασίες της Επιτροπής ΠΑΝΑ κάτι το οποίο μας βοηθά πολύ, γνωρίζετε τα προβλήματα που υπάρχουν και είναι καλό να συνδέσουμε τα θέματα αυτά και με τις υπόλοιπες διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίσουμε εμείς τον προϋπολογισμό από τη μία και τη φορολογία από την άλλη οι πολίτες δεν θα καταλάβαιναν να τους προετοιμάζουμε για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και των νέων τεχνολογιών και από την άλλη να εξακολουθούμε να, κάνουμε, να χάνουμε φόρους από τον προϋπολογισμό. Πάντως δύο θέματα πρέπει να φωτιστούν. Πρώτον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει ένα προσανατολισμό δημοσιονομικό συνολικά ουδέτερο για το σύνολο της ζώνης ευρώ η ανάπτυξη έχει λιγότερη ε, ανάγκη από οικονομική στήριξη αλλά από την άλλη θα ήταν πρόωρο να πούμε ότι δεν τη χρειαζόμαστε καθόλου. Από την άλλη προτείνουμε πολιτικές οι οποίες ε, στηρίζουν την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Εσείς υπογραμμίσατε τη σημασία αυτής της διάστασης στις προηγούμενες εκθέσεις σας. Εμείς έχουμε κάποιες συστάσεις οι οποίες ποικίλουν ανά φυσικά και ζητάμε από όλα τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα ευνοήσουν την δημιουργία θέσεων απασχόλησης ποιότητας που να βασίζονται στις ανάγκες βέβαια της αγοράς εργασίας. Εμεί ζητάμε από τις χώρες οι οποίες έχουν ένα έλλειμμα τρεχουσών πληρωμών ή ένα υψηλό χρέος εξωτερικό να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Κανένας δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από μια κατάσταση τέτοιου επίπεδου. Και ζητάμε από τις χώρες επίσης οι οποίες έχουν υψηλά πλεονάσματα να βοηθήσουν την αύξηση των μισθών και να δώσουν κίνητρα στην ε, εσωτερική ζήτηση. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι η ανάπτυξη αυτή, η υψηλότερη εδώ και 10 χρόνια, να ωφελήσει όλους και αυτούς οι οποίοι έχουν ένα υψηλό χρέος να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουν να επενδύσουν και αυτοί που έχουν ένα περιθώριο με τα πλεονάσματα να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν τις επενδύσεις υπέρ των πολιτών τους. Μπορούμε να επανέλθουμε στις προκλήσεις αυτής και στη συνέχεια των συζητήσεών μας σχετικά με τις νομοδοτήσεις για τα σχέδια των προϋπολογισμών αλλά προς το παρόν θα μείνω σε αυτά τα γενικά που σας είπα και είμαι όπως και ο Βάλντι στη διάθεσή σας ε, για ερωτήσεις στις οποίες ίσως μπορούμε να απαντήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε και τους δύο για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Τήρησατε επίση και το χρονικό όριο. Λοιπόν, στον πρώτο γύρο, στους δύο εισηγητές από την Econ και την Έμπλη για το θέμα της ετήσιας έκθεσης πρόοδου. Είχαμε εισηγητή από τους Ελληνικούς Δημοκρατές, αλλά δυστυχώς ο κύριος Βάιρ δεν είναι εδώ, είναι στο νοσοκομείο, αλλά έχουμε ε, τον συνάδελφο Περέιρα. Έχετε τρία λεπτά παρακαλώ για τα σχόλια και ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να καλωσορίσουμε και τους ε, δύο επιτρόπους εξ ονόματο του εισηγητή και της ομάδα μας να πούμε ότι αρχικά αυτός ο διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής είναι πολύ σημαντικός ε, για ένα πιο δημοκρατικό ευρωπαϊκό εξάμεινο και έτσι και μια πιο ε, δημοκρατική οικονομική και δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωζώνη. Με τα χαράς ε, βλέπουμε βελτίωση στις οικονομικές επιδόσεις και αναγνωρίζουμε ότι το λεγόμενο τρίγωνο των επενδύσεων, των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων και της υπεύθυνη δημοσιονομικής πολιτικής ε, φέρει καρπούς, από ό,τι φαίνεται. Ωστόσο, θέλουμε να επισημάνουμε ότι είναι θετικό που στην ανακοίνωσή σας υπάρχει αναφορά στην ανάγκη επιπρόσθετων μέτρων ε, για να διευκολύνουμε ε, τις επενδύσεις και να αυξήσουμε το, τα οικονομικά αποτελέσματα. Ε, η υπερβολική εξάρτηση από την οικονομική πολιτική δεν επαρκεί. Αντιθέτως, πρέπει να αναμένουμε αλλαγές στη δημοσιονομική και νομισματική μάλλον πολιτική στο προσοχές μέλλον. Οπότε χρειαζόμαστε και μια καλύτερη στήριξη από τη δημοσιονομική πολιτική. Δεν είμαι βέβαια όμως ότι η έκθεση προόδου που μας παρουσιάσατε ακολουθεί αυτά τα επίπεδα φιλοδοξιών. Ιδίω, επειδή η ετήσια έκθεση προόδου προτείνει μια ε, σφαιρικά ουδέτερη δημοσιονομική στάση, φορολογική στάση για το 2018. Ε, νομίζω ότι αυτή η πρόταση προκαλεί έκπληξη και απογοήτευση ε, έκπληξη γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι είχε προτείνει το αντίθετο. Μία ε, κατά κάποιον τρόπο επεκτατική, ε, μετριοπαθή επεκτατική πολιτική. Γιατί υπάρχει χαμηλή ανάκαμψη Επιπλέον, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει σε ε, ποσοτικούς ε, αριθμούς το, την ανάγκη παρέμβασης για το 2017. Οπότε αναρωτιόμαι κατά πόσο η αλλαγή στην οικονομική κατάσταση είναι τόσο σημαντική για να εξηγήσει μια τέτοια μεταβολή στην πολιτική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία τώρα καλεί μία ε, ουδέτερη στάση, παρότι ξέρουμε ότι είχαμε μια τέτοια ε, στάση για το 2017 και το 2018. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι επιστατικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει και πάλι οι χώρες που έχουν το περιθώριο να κάνουν περισσότερα, να επενδύουν, να συμβάλλουν ε, στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, όμω από ό,τι φαίνεται ε, εκείνες δεν ακούνε. Οπότε να ρωτήσω τους επιτρόπους τι μπορούν να κάνουν και τι θα κάνουν προκειμένου αυτή η σύσταση που είναι τόσο σημαντική για την ε, οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης να γίνει ακουστή. Ευχαριστούμε πολύ. Από πλευρά Σέμπλ τώρα, ο κύριος Κρίστοφ Χέτμαν από το ΕΛΚ. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, αξιότιμη Επιτροπή, έχουμε δει την έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρκετά θετική. Υπάρχει οικονομική ανάκαμψη και από ό,τι φαίνεται αυτό διατηρείται ως τάση και συνοδεύεται και από χαμηλότερη απασχόληση και χαμηλότερους, ε, υψηλότερη απασχόληση, μάλλον και χαμηλότερους δείκτες ε, φτώχειας. Όμως αυτό δεν ισχύει σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν κάποια στοιχεία κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης που είναι πολύ ενθαρρυντικά παρότι η ενεργεία των νέων ε, διατηρείται σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα και θα πρέπει να είναι από τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των κρατών μελών μέσα στην επόμενη χρονιά. Με τα χαρά βλέπουμε περισσότερου πόρου για την απασχόληση των νέων και τη σχετική πρωτοβουλία. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ θα στηρίξει τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την ε, τροποποίηση των εκπαιδευτικών του συστημάτων και την προσαρμογή του ε, προ την αγορά εργασία. Υπάρχει ένα έλλειμμα σε τη φορά τις ψηφιακές δεξιότητες. Γι' αυτό ίσως να έχουμε και υψηλά επίπεδα ανεργίας στους νέους. Παρότι υπάρχουν πολλές ε, κενές θέσεις εργασίας ε, στην οικονομία. Και ακόμα ένα ερώτημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Μα το αναφέρουν και επιχειρηματίε που θεωρούν ότι αυτό είναι σημαντικό φραγμό προ την ανάπτυξη. Όμω υπάρχουν ε, άλλες περιοχές και άλλοι τομεί όπου η ε, ανεργία είναι απαράδεκτα υψηλή. Ποιο είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτήν την κατάσταση και πώ μπορεί να στηρίξει και τι δύο πλευρέ και να τους ενθαρρύνει να αξιοποιούν άλλα εργαλεία πέραν των τεντρημένων βλέπουμε ότι σε ό,τι αφορά την αγορά εργασία, αυτή τη στιγμή δεν μιλούμε μόνο για την ε, αγορά εργασία του εργοδότη, αλλά και του εργαζομένου. Για να μειώσουμε την ανεργία χρειαζόμαστε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις και να άρουμε όλους τους φραγμούς για την ε, δημιουργία θέσεων εργασίας. Να στηρίξουμε τις νέες τεχνολογίες γιατί έχουν πολύ σημαντική δυναμική σε ό,τι αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων. Θεωρώ ότι όχι μόνο το ΕΦΣΙ αλλά και τα διαθροτικά ταμεία και άλλα είδη επενδυτικών ταμείων θα πρέπει να αξιοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση γιατί έχει ήδη αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά τους ε, στην στήριξη των επενδύσεων αυτών που θα ε, κλείσουν αυτό το, το χάσμα, θα γεφυρώσουν αυτό το χάσμα ε, των ανισοτήτων. Σημαντική είναι και η γεωγραφική διάσταση και η γεωγραφική ανισομέρεια μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μια ολιστική σφαιρική προσέγγιση, γιατί βέβαια θέλουμε να ενθαρρύνουμε ε, του ε, εργαζόμενου να συμμετάσχουν στην αγορά εργασία. Όμω χρειάζεται γι' αυτό μια στοχοθετημένη κοινωνική πολιτική που διασφαλίζει μια ισορροπία μεταξύ του επαγγελματικού και του οικογενειακού του βίου. Επομένως, ε, καλό είναι να αξιοποιούνται διάφορες μορφές ε, ελαστικής ε, απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης και διαμόρφωσης νέων υποδομών. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλές, πολλές είναι ευκαιρίες από τις εταιρικές σχέσεις δημόσιο-δυτικού τομέα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δομπρόφσκης πρώτα να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ ε, για τα ερωτήματα που θίξατε. Πρώτον, ε, για τις ε, συνολικές προτεραιότητες πολιτικής, πράγματι εκτιμούμε ότι χρειαζόμαστε όλα αυτά τα στοιχεία, τι επενδύσει, τι δυτικέ μεταρρυθμίσει και τη δημοσιονομική πολιτική. Αυτό το τρίγωνο λοιπόν ε, ε, ε, φέρει αποτελέσματα, όμως οι επενδύσεις ανακάπτουν μόνο τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, οπότε απαιτείται ακόμα πολλή δουλειά για να ενισχύσουμε αυτές τις επενδυτικές τάσεις. Και αυτές τις πρωτοβουλίες φάνηκαν και από το ΕΦΣΥ, αλλά επιβεβαιώνω και ότι τα ευρωπαϊκά διασωτικά και επενδυτικά ταμεία διδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση και την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και για τη βελτίωση του ε, επιχειρηματικού περιβάλλοντος για να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα την νομισματική πολιτική και την Ευρωζώνη, για τη δημοσιονομική στάση στην Ευρωζώνη, Πράγματι, αυτή τη στιγμή συνιστούμε μία ε, γενικώς ε, ουδέτερη και ισορροπημένη ε, δημοσιονομική στάση για να διασφαλίσουμε και την ανάπτυξη αλλά και την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, ιδίως ε, για τις χώρες που έχουν υψηλά επίπεδα ε, χρέους και λύματο, για να τα φέρουμε όλα αυτά κάτω λοιπόν, να τα περιορίσουμε. Και αυτή ήταν και συζήτηση πέρσι κατά πόσο ε, μία μετριοπαθώς επεκτατική δημοσιονομική στάση είναι πλέον κατάλληλη. Πρέπει να πούμε όμως ότι η οικονομική ανάκαμψη συνεχίζεται και ενισχύεται μάλιστα. Πρόσφατα ε, αναβαθμίσαμε τις οικονομικές μας προβλέψεις προς τα πάνω και τις αναθεωρήσαμε προς τα πάνω. Οπότε μια γενικά ουδέτερη ε, δημοσιονομική στάση θεωρούμε ότι είναι πλέον κατάλληλη και ισορροπημένη και αυτή τη γνώμη συμμερίζεται και το ε, Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο που συστάθηκε πρόσφατα. Τώρα για τα ερωτήματα που θίξατε για τη στήριξη της απασχόλησης, ιδίως για την απασχόληση των νέων. Μία από τις ε, πρώτες προτεραιότητε ε, της ε, Επιτροπή αυτής, η παροχή μεγαλύτερη στηρίξη για την πρωτοβουλία για τους νέους και την εγγύηση της νεολαίας. Θέλουμε να ενισχύσουμε τους συνδέσμους μεταξύ αγοράς, εργασίας και εκπαιδευτικών συστημάτων. Αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε με το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων. Να διασφαλίσουμε ότι ε, τα αποτελέσματα της, ε, του εκπαιδευτικού συστήματος, ιδίως της επαγγελματικής κατάρτισης, καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε δυτικά για να ε, υλοποιήσουμε τις επιμέρους πρωτοβουλίες του θεματολογίου μας για τις δεξιότητες. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε και μια εβδομάδα δεξιοτήτων όπου συζητήσαμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και λύσεις και προτάσεις για το μέλλον. Τώρα, αναντιστοιχεία μεταξύ ανεργίας και προσφοράς εργατικού δυναμικού. Υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα είναι δομικό και εδώ ε, αυτό θέλουμε να λύσουμε με το θεματολόγιο δεξιοτήτων. Και το άλλο είναι γεωγραφικό. Υπάρχουν συζητήσεις και για την κινητικότητα των εργαζομένων αλλά βέβαια όταν εξετάζουμε τέτοια θέματα πρέπει να έχουμε κατά νου παράγοντες όπως είναι η διορία εγκεφάλων, η φυγή των νέων προς ξένες χώρες, γιατί όταν ε, άνθρωποι με δεξιότητες και νέοι ε, φεύγουν από τις χώρες τους, αυτό τελικά δημιουργεί πρόβλημα σε αυτές τις χώρες και περιφέρειες. Και μένω εδώ. Uh, Ο Επίτροπος Επανέλθομαι σε αυτά τα οποία είπατε στο, στην προηγούμενη σειρά. Πράγματι τα πράγματα άλλαξαν από πέρυσι. Πέρυσι είχε κρυθεί αναμένο να στηριχθεί η ανάπτυξη γιατί θεωρείται ιδιαίτερα άνηση και ιδιαίτερα εύθραυστη και γι' αυτό θελήσαμε μέσω μιας σημαντικής δημοσιονομικής στήριξης να βοηθήσουμε και γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει, πρότεινε για πρώτη φορά μετά από καιρό μια θετική τάση. Η παρατήρηση αυτή είχε γίνει δεκτή και από το Eurogroup και από το Συμβούλιο και τέλος αναφέρθηκε πλέον σε μια ουδέτερη δημοσιονομική πρόταση. Και είχαμε δίκιο γιατί το συνολικό τελικά αποτέλεσμα ήταν ελάχιστα θετικό το 2017. Είναι ελάχιστα θετικό για το 2017. Και γι' αυτό έχει υπάρξει και αυτή η ισχυρή ανάπτυξη, ισχυρότερη από τις αναλύσεις μας. Πράγματι λοιπόν πιστεύουμε ότι τώρα πια η ανάπτυξη δεν χρειάζεται πλέον τόση δημοσιονομική στήριξη αλλά ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμα και τώρα ανάγκη ενίσχυση της ανάπτυξης. Δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια, φάση, σε ποια του κύκλου ανάπτυξης βρισκόμαστε και γι' αυτό κάποια στήριξη απαιτείται. Και γι' αυτό ε, έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι αυτή η ουδέτερη αν θέλετε προοπτική είναι αυτό το οποίο θα ζητήσουμε και θα προτείνουμε στο Συμβούλιο και ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα δεχθεί την πρόταση αυτή γιατί πράγματι νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Ένα δεύτερο σημείο αναφέρεται σε αυτά τα οποία μας είπατε για τις χώρες ε, οι οποίες έχουν σημαντικότατα πλεονάσματα και χώρες αυτές δεν θεωρείται ότι πρέπει να, ε, να κάνουν δεκτές τις προτάσεις μας σχετικά με τη διάθεση του πλεονάσματος σε επενδύσεις έχετε σχεδόν δίκιο. Στην Γερμανία γίνεται μια μεγάλη συζήτηση και υπάρχουν κάποιες εξελίξεις προς την κατεύθυνση των επενδύσεων αλλά απαιτούνται να γίνουν περισσότερα. Εμείς αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι για μια ακόμη φορά να θέσουμε τη συζήτηση αυτή στο Eurogroup Νομίζω ότι και οι δικές σας συστάσεις και οι δικές σας πιέσεις έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο και θα συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε την ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις και σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο του ιδιωτικού τομέα έτσι ώστε και αυτές οι χώρες με το ισχυρό πλεόνασμα να μπορέσουν να καλύψουν το κενό επενδύσεων που μπορεί να υπάρχει και να αναπτυχθεί συνολικά και η Ευρωζώνη. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στην Γερμανία πλέον, ξέρουμε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για το σχηματισμό της κυβέρνησης συνασπισμού. Ελπίζω να έχουμε σύντομα μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση, κάτι το οποίο θα βοηθήσει την ενίσχυση των επενδύσεων. Εμείς θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε την κατάσταση στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στον δεύτερο γύρο τους σκιώδεις εισηγητές και τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. 1,5 λεπτό ο καθένας. Ακούσαμε στην αρχή από τους σοσιαλιστές το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το ECR. Τώρα έχει το λόγο η Άγνες Σογκάριος. Λέει η Επιτροπή ότι θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από την ανάπτυξη εκ νέου της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρώπη και έχει σημασία ότι θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση από μια θετική νότα. Έχει επίσης σημασία να πούμε ότι η ανάπτυξη, η ανάκαμψη καλύτερα γίνεται με πολύ άνισο τρόπο. Η κατανομή ε, των κερδών αν θέλετε, των ωφελημάτων δυστυχώς είναι άνηση και πάντα υπάρχουν ισχυρά επίπεδα φτώχειας και πρέπει εδώ να στρέψουμε την προσοχή μας. Εσείς ο ίδιος αναφερθήκατε στα χαμηλά επίπεδα ανάκαμψης των αμοιβών σε αυτούς που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και στην κοινωνική προστασία και τη χειροτέρευση των συνθήκων εργασίας. Έγινε όμως τώρα η συνάντηση στο Χέτεμπορκ και αυτά τα επιπλέον μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσουν. Βέβαια μια διακήρυξη παραμένει ε, ισχυρή σε συμβολικό επίπεδο και μετά τη διακήρυξη θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα μέτρα ιδιαίτερα στις ανισότητες στην απασχόληση κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό δυστυχώς σε πολλές χώρες. Μία ερώτηση να κάνω τώρα για τον κοινωνικό διάλογο και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας των εργαζομένων. Και συνάδελφοι, ένα πράγμα είναι να λέει κανείς ότι διεκδικώ μια αύξηση. Από την άλλη όμως όταν έχει συρρυκνωθεί τόσο πολύ και συμπιεστεί τόσο πολύ η διαπραγματευτική μας ικανότητα, πώς μπορούμε να ελπίζουμε σε αυξήσεις αμοιβών, ακόμα και σε χώρες όπως οι κάτω χώρες και η Γερμανία γιατί μιλάμε για χώρες που ναι μεν αναπτύσσονται με υψηλούς ρυθμούς αλλά δυστυχώς οι μισθοί ε, καταραίουν ουσιαστικά ακόμα και στις χώρες με υψηλά πλεονάσματα. Από τον και το Έλικο, ο κύριος Χόκμαρκ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση που μας κάνατε και νομίζω ότι όλοι καλωσορίζουμε το γεγονό ότι πολλά από τα αριθματικά στοιχεία είναι αρκετά ευνοϊκά στην παρούσα φάση. Να ευχαριστώ σε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, έφτασε το θέμα τη ε, ουδέτερη δημοσιονομική συστάσης και το ζητήσαμε αυτό από πλευρά Κοινοβουλίου την τελευταία φορά και συζητούσαμε πώ θα το πετύχουμε μάλιστα αυτό. Να επανέλθω όμω αν μου επιτρέπετε, σε μία από τι προτάσει που περιλαμβάνονται και στην ετήσια έκθεση ανάπτυξη. Πραγματικά πάρα πολύ βασική και κρίσιμη σημασία στην εισαγωγή αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει επιπλέον ε, τα ποσοστά ΑΕΠ και παραγωγικότητας παραμένουν κάτω από το ε, βέλτιστο επίπεδο και τα επίπεδα ε, επενδύσεων είναι κάτω από το ποσοστό που ήταν πριν από την κρίση. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μα το γεγονό ότι οι επενδυτέ είναι ακόμα διστακτικοί, πιο διστακτικοί από ότι πριν από την κρίση, αποτελεί το πιο δύσκολο, αν θέλετε, κομμάτι των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Αν αυτό δεν το αντιμετωπίσουμε, ούτε καινοτομία θα έχουμε επαρκή, ούτε ανταγωνιστικότητα, ούτε ποσοστό παραγωγικότητα. Αυτό που μου προκαλεί λοιπόν έκπληξη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για το πώς θα διευκολύνει τις επενδύσεις αυτές, δεν μιλάει τόσο πολύ για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονομία της θα καταστεί πιο ελκυστική για τους επενδυτές. Υπάρχει ένα πλεόνασμα τέτοιων επενδύσεων στην Ευρώπη. Δεν τις προσελκύουμε όμως. Αυτό είναι θέμα κρατών μελών και πολλά άλλα τέτοια ζητήματα από αυτά που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εξαρτάται προφανώ και από τι μεταρρυθμίσει επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε μα, σα παρακαλώ, πώ θα επίλυσετε αυτό το θεμελιώδε πρόβλημα. Ευχαριστώ, Κούναρ. Από το ECR εκπροσωπούνται και οι δύο επιτροπέ από την κυρία Τρεμπέσιου, η οποία και έχει τρία λεπτά, αν το επιθυμεί. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς κύριε Επίτροπη που ήρθατε εδώ. Αναφερθήκατε σε πολλά αριθμητικά στοιχεία, σε πολλούς αριθμούς. Για να γίνει όμως μια σωστή οικονομική ανάλυση χρειάζονται και σωστά αριθμητικά στοιχεία και αυτό είναι επικίνδυνο στην παρούσα φάση το να βρούμε σωστά αριθμητικά στοιχεία γιατί στην Ελλάδα ο πρώην πρόεδρος ε, επικεφαλής ε, της στατιστικής υπηρεσίας ε, καταδικάστηκε σε μεγάλο πρόστιμο 10.000 ευρώ γιατί, βελτί... γιατί διόρθωσε τα απατηλά στοιχεία που είχαν χορηγήσει οι προκάτοχοί του. Και ο Χατζηγεωργίου λοιπόν, ο οποίος τα αποκάλυψε όλα αυτά, ε, κατηγορείται. Το ερώτημα λοιπόν που σας απευθύνει το εξή θα αναμειχθείτε εδώ, γιατί δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ιστορικό θέμα της Ελλάδος. Όταν διορθώνονται δηλαδή εσφαλμένα στατιστικά στοιχεία Ιδιαίτερα όταν είναι κάνει σε μια νομισματική ένωση, είτε πρόκειται για Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είτε για άλλο θεσμικό όργανο, θα πρέπει να μπορούμε να θεωρούμε ότι είναι σωστά τα στοιχεία. Μία άλλη ερώτηση. Έχουμε παραπονηθεί έχετε παραπονηθεί μάλλον για το γεγονός ότι η Γερμανία, η χώρα μου, είναι πάρα πολύ δυνατή, υποτίθεται, αλλά μήπως θα πρέπει να κοιτάξουμε και γίνεται με την Ιταλία. με υψηλή χρέωση, με μη εξυπηρετούμενα δανεί και βλέπουμε λοιπόν ότι στη χώρα αυτή η σύγκληση την οποία αναφέρεται δεν υπάρχει. Η ανάπτυξη μεταξύ των χωρών είναι πολύ διαφορετική. Και μια τελευταία ερώτηση επιτρέψτε μου για το πρεστή τη Τρέχουσα επιτροπή, ό,τι αφορά την πρωτοβουλία κατά της ανεργία των νέων. 500 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται ω τώρα για το έργο αυτό. Τα μισά εξ αυτών έχουν ε, δαπανηθεί στην παρούσα φάση. Με τους πόρου λοιπόν αυτούς, με τα κονδύλια αυτά, ε, έχουμε βοηθήσει την Ισπανία και την Πορτογαλία κυρίω. Ε, αλλά υπήρξε δυσκολία απορρόφησης από τις χώρες αυτές μέσω των κρατικών δημόσιων δομών. Η Ισπανία όμως και η Πορτογαλία είναι αυτές οι χώρες που έχουν καλά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ενεργείας των νέων. Άρα η επιτυχία έχει να κάνει πιο πολύ με τις χώρες της ίδιας παρά με το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για πείτε μας λοιπόν, πώς εξηγείται αυτή την απόκληση των στοιχείων. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και θα ήθελα τώρα να στραφώ πάλι προ τον Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κ. Ντόμποφσκη, και πάλι 8 λεπτά συνολικά έχετε το λόγο παρακαλώ για απαντήσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, άκουσα πολλέ ερωτήσει. Καταρχά. Όντω. σε ό,τι αφορά την ανάκαμψη, ναι, υπάρχει η ανάπτυξη, αλλά είναι άνηση ακόμα. Άνηση ανάπτυξη. Συζητάμε λοιπόν την αιτήσια ανάπτυξη και θέτουμε προτεραιότητε και φέτο και τα τελευταία χρόνια. Και φέτο λοιπόν δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ε, συμπεριπτική αυτή ανάπτυξη. Ανάπτυξη για όλους. οικονομική ανάπτυξη να φτάσει σε όλους, ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους από τι κοινωνίε μας. Και αυτή η προσέγγιση αποτυπώνεται στις συστάσεις αναχώρα τις οποίες θα υποβάλουμε προς τα κράτη. σκοπεύουμε να το κάνουμε και στις συστάσεις αναχώρα για του χρόνου. Ακούσαμε τώρα τον ότι ο αντίκτυπος του κοινωνικού πυλώνα για το ευρωπαϊκό εξάμεινο ε, είναι ιδιαίτερος. Όπως σας είπαμε και στη Σύνοδο, σκοπός μας τώρα είναι να ληφθούν υπόψη ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων και γι' αυτό η κοινή έκταση απασχόλησης φέτος αναφέρει το νέο κοινωνικό scoreboard των πίνακα επιδόσεων. Θα υπάρχει καταμέτρηση λοιπόν των εθνικών μεταρρυθμίσεων στο τέλος του πίνακα αυτού και σε ό,τι αφορά τις φιλοδοξίες που έχουν ε, οριστεί στον πυλώνα. Σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό διάλογο και την ε, δυνατότητα διαπραγμάτευσης Πρόκειται για ένα από τα θέματα τα οποία θα ακολουθήσουν, που ακολουθούμε συγγνώμη πάρα πολύ στενά σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό διάλογο στα κρατημέλη. Και πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τον κοινωνικό διάλογο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του δυναμικού των κοινωνικών εταίρων και λοιπές πρωτοβουλίες μεταξύ των οποίων και η υποστήριξη ε, του ρόλου των ε, ε, κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Στη συνέχεια, το θέμα της παραγωγικότητας και των επενδύσεων. Αυτό το θέμα της παραγωγικότητας το υπογραμμίζω και το υπογράμμισα και στα εισαγωγικά μου σχόλια. Γιατί πραγματικά θέλουμε να αυξήσουμε την ευημερία σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Χρειάζεται λοιπόν αναπτυσσόμενη παραγωγικότητα. Για αυτή με τη σειρά τη προαπαιτούνται επενδύσει. Και γι' αυτό λοιπόν μία από τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτο ήταν το σχέδιο επενδύσεων για την Ευρώπη, το σχέδιο Juncker και το το στρατηγικό ταμείο, το ταμείο στρατηγικών επενδύσεων και βλέπουμε ότι αυτό έχει σκοπό να προωθήσει τις επενδύσεις και πραγματικά θα πρέπει να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει και μια διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, γι' αυτό προβαίνουμε και στις συστάσεις αναχώρα Προς τα κράτη-μέλη, ακριβώς για το θέμα αυτό, το περιβάλλον των επιχειρήσεων. Κάποιες από τις ερωτήσεις τώρα που ακούσαμε, πιο συγκεκριμένα για τις μεμονωμένες χώρες, για την ε, Ελλάδα και την Στατιστική Υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σαφώς τοποθετηθεί και έχει εκφράσει ανησυχίες. Φυσικά θα πρέπει να σεβαστούμε την ανεξαρτησία των εθνικών δικαστικών συστημάτων, αλλά όντως αληθεύει επίσης ότι τα κρατή-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν και να έχουν ε, ανεξάρτητα και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Διαπιστώνουμε λοιπόν από την κρίση και μετά από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα όσα έχουμε δει μας ε, προκαλούν ε, απόλυτη εμπιστοσύνη στα στατιστικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ανεξαρτησία των στατιστικών υπηρεσιών, γιατί αυτό είναι στον πυρήνα, αν θέλετε, ε, της διαδικασίας και στον τομέα της Ευρωζώνης. Στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να πω ότι η Ιταλία δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει τα υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Έχουμε κι άλλες. Και γι' αυτό στην παρούσα φάση καταρτίζουμε μια στρατηγική για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Η πρωτοβουλία για την ανεργία των νέων. Φυσικά υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα εκείνα όπου έχουν υψηλή ανεργία των νέων. Και φυσικά δεν είναι όλα ξεκάθαρα και απλά, αλλά σημειώνουμε πρόοδο θα έλεγα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της πρωτοβουλίας ε, για την ανεργία των νέων, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία. Ευχαριστώ πολύ, ο κ. Μοσκοβισή. So, ε, briefly. Πολύ σύντομα, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις επενδύσεις για να απαντήσω το προηγούμενο σχόλιο. Νομίζω αρχικά ότι οι προβλέψεις επένδυσης, ανάπτυξης μάλλον, βοηθούν και θα πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με τα ε, μικροοικονομικά. Πράγματι, πρέπει η Ευρώπη και είναι πιο ελκυστική η Ευρώπη πλέον, αλλιώς θα είχαμε τέτοια αποτελέσματα. Ωστόσο, και έχετε δίκιο, πρέπει να επιμείνουμε στις δικές μεταρρυθμίσει στα κράτη-μέλη. Όχι επειδή δηλαδή, τα πράγματα πάνε καλύτερα ξαφνικά να εγκαταλείψουμε αυτή τη φιλοδοξία ε, μεταρρύθμιση της οικονομίας μας. Αντιθέτως, πολύ καλό που έχουμε βγει από την κρίση, αλλά πρέπει πάντα να αποτρέψουμε και την επανάληψη ε, τέτοιων φαινομένων στο μέλλον. Και εμένα στον τρίτο πυλώνα του προγράμματος Juncker, που έχει να κάνει με τις επενδύσεις. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι μία ε, σημαντική προώθος. Και αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να ακολουθούμε για να έχουμε μια καλή ε, προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Για τα στατιστικά στοιχεία στην Ελλάδα. Είναι ένα λεπτό ζήτημα. Πραγματικά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αφενός, η τρέχουσα επιτροπή πάντα αναγνωρίζει και δέχεται τα στοιχεία που μας ε, έδωσε αυτό το πρόσωπο στο παρελθόν για τα δημοσιονομικά στοιχεία της Ελλάδας. Από την άλλη μας ζήτησαν από το Υπουργείο Οικονομικών αυτή η κατάσταση που γενικά είναι άδικη να επιληθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Και στη συζητήση μας, στο πλαίσιο και της εξέτασης του ελληνικού προγράμματος με τους ομολόγους μας, με τον Υπουργό κ. Τσακαλώτο, έχουμε θίξει πολλές φορές αυτό το ζήτημα ε, και το έχουμε κάνει και δημοσίως. Οπότε η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ιδιαίτερα γνωστή και από ό,τι κατάλαβα καλά συμφωνείτε κι εσείς. Όμως γνωρίζουμε όλοι ότι ε, τις χώρες μας διέπει το κράτος δικαίου, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και έτσι δεν μπορούμε να το παρακάνουμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην ε, διατρέχουμε τον κίνδυνο παρεμβολής στην δικαστική διαδικασία. Γι' αυτό και μπορούμε μόνο να επαναλάβουμε τη δική μας θέση. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια κοινή συνεδρίαση αυτή της ε, Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και τη Επιτροπής Απασχόλησης. Να δώσω το λόγο στην Μαρίτα Λούσκοφ, ε, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής ΕΜΠΛ, που θα προεδρεύσει του δεύτερου τμήματο ε, τη συνεδρίασης. Ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν στον τρίτο γύρο. Ο κάθε μιλητή έχει 1,5 λεπτό στην διαθεσή του. Ξεκινούμε με μέλος της ΕΚΟΝ, Καρολίνα κάλα από την Άλντα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή αναφέρει ότι η γενοτομία και η ανταγωνιστικότητα είναι σημαντικά στοιχεία και ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να βελτιώσουν τι αγορέ του στο μέλλον. Συμφωνώ απολύτω και φαντάζομαι όλοι εδώ συμφωνούν. Αν δείτε την καινοτομία ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική ε, ανισότητα στις επιδόσεις ε, των κρατών μελών. Οι επιδόσεις στη καινοτομία πάνε χέρι-χέρι με την θέση ανταγωνιστικότητας του κάθε κράτους μέλους. Κάποιες χώρες συνεχώς υπολείπονται των υπολείπων σε ό,τι φορά καινοτομία και ως εκ του και ε, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα. Οπότε, τι συγκεκριμένες δράσεις μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει τις ε, χώρες ε, ουραγούς να επιταχύνουν και να τα πάνε καλύτερα. Και δεύτερον, κάποιες από αυτές τις χώρες που υπολείπονται στον τομέα της καινοτομίας είναι και οι χώρες που οι πλέον υπερχρεωμένες και αυτές είναι μάλλον οι χώρες που επενδύουν περισσότερο, μάλλον αξιοποιούν μεγαλύτερο τμήμα του προπολογισμού για να καλύψουν τρύπε παρά για να επενδύσουν στο μέλλον. Τι θα κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι οι προπολογισμοί των κρατών μελών θα έχουν μία σύνθεση πιο φιλική προ την ανάπτυξη. Θεωρείτε ότι έχετε κάνει αρκετά ω προ αυτή την άποψη. Ευχαριστώ. Καλπέσα μου από την άλλη επίση, από την Επιτροπή Απασχόλησης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά για να με καταλάβει καλύτερα ο κύριος Μοσχοβησή, τον οποίο χαιρετώ, όπως και τον κύριο Ντομπρόσκης φυσικά. Στον τομέα της απασχόλησης ε, και της κοινωνικής πολιτικής η παρέμβαση μου ακολουθεί ακριβώς τη συνάντηση κορυφής του Χέτεμπερ και γι' αυτό στα πλαίσια αυτά θα ήθελα να αναφέρω ότι πήρα άλλωστε μέρος και στον τομέα της απασχόλησης στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θέτει δύο προϋποθέσεις. Από τη μία δημιουργία νέων θέσεων με ποιότητα φυσικά και ε, δεύτερον ε, οι ανισότητες οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν και που ε, πράγματι κάνουν την κοινωνία μας να τρέμει. Πρέπει λοιπόν να αντιδράσετε. Υποτίθεται ότι έχουμε ξεφύγει από την χρηματοπιστωτική κρίση, θυμίζω. Οπότε τίθενται ακόμα και τώρα πάρα πολλά θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις της θα λάβει άραγε υπόψη αυτήν την αυξανόμενη ανισότητα ανάμεσα στις κοινωνικές κατηγορίες. Το θέμα το οποίο δημιουργείται σε κοινωνικό επίπεδο είναι κάτι το οποίο θα είναι στο μέλλον καθοριστικό για την υιοθέτηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Μπορούμε να έχουμε, εν πάση περιπτώσει, μια ανάπτυξη στραμμένη στη συνοχή. Σας ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος της ΓΟΥ έχει το λόγο, Μιγγέλ έχει το λόγο. Η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σημειώνουν πάρα πολλά προβλήματα έλλειψης επενδυτικών δυνατοτήτων στην Ευρώπη. Η έκθεση αυτή μας επιτρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν φτάσει στα επίπεδα που είχαν πριν την κρίση. Αλλά οι δημόσιες επενδύσεις είναι στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 20 χρόνια, 0,2% ιδιαίτερα στις υποδομές. Ο λόγος είναι προφανής, είναι το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και οι πολιτικές λιτότητας που επιβάλλονται στα κράτη-μέλη, πολιτικές οι οποίες είναι αποκλειστικά δημοσιονομικές. Ακόμα και ο Υπουργός Μοντόρο στη χώρα μου πήρε μέρο στις συζητήσει για να αποτρέψει αυξήσεις δαπανών στον τομέα των κοινωνικών και στον τομέα των υποδομών. Τη στιγμή λοιπόν που εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε επενδύσεις χωρίς εμπόδια, μήπως θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε και το σύμφωνο σταθερότητα το οποίο είναι το βασικό εμπόδιο για τις δημόσιες επενδύσεις σήμερα. Και μια δεύτερη ερώτηση. Αν μια χώρα ζητήσει να μην υπακούσει στην ρήτρα ευελιξίας στον τομέα των υποδομών μέσω δημοσίων επενδύσεων. Τι θα απαντήσετε κύριε Μοσκόβηση. Η κυρία Κούνεβα έχει το λόγο. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί κύριε Επίτροποι, η ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη που μας παρουσιάσετε είναι γεμάτη από θριαμβευτικές δηλώσεις για την απασχόληση. Σημειώνεται πως η ανεργία βρίσκεται στα πιο χαμηλά ποσοστά από το 2018, 7,6 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 9,1 στη ζώνη του ευρώ. Καταρχάς, δεν είναι ανησυχητικό πως η ζώνη του ευρώ έχει μεγαλύτερη ανεργία είδατε πόσο υψηλά είναι τα ποσοστά σε Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα. Και έχουμε αναρωτηθεί για τι θέσει εργασία πρόκειται. Σε συντεδεμένη έκθεση για την απασχόληση σημειώνεται πω μόνο το 14% των θέσεων εργασία είναι μόνιμε. Χαίρομαι πάντως που μιλάτε για ενεργητικέ πολιτικέ απασχόληση ειδικά για πώ μακροχρόνια άνεργους και τους νέους η αξιοποίηση του πακέτου Juncker διότι έξι υπουργοί απασχόληση Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ελλάδα, ακριβώ λόγω τη ανησυχητικών τάσεων που εμφανίζονται ω μόνιμε σε αυτέ τι κατηγορίε εργαζομένων υποβάλλουν μια διπλή πρόταση για τις χώρες της ανεργία υψηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η πρώτη, τουλάχιστον το 5% του πακέτου Juncker να παρουσιάζεται για κονδύλια πολιτικών απασχόληση με δυνατότητα συγχρηματοδότησης και πάνω από 50% μέτρο που έχει εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις. Και δεύτερο, οι πόροι που θα διαθέτονται για προγράμματα απασχόληση, τα οποία στηρίζει ω μοχλό ανάπτυξη η έκθεση να εξαιρούνται από τον υπολογισμό των δίκτων, του Σύμφωνου σταθερότητα. Η πρόταση αυτή θα παρουσιαστεί σύντομα τόσο σε εσά όσο και στον κύριο Γιούρκεν και στηρίζεται ήδη από 32 βουλευτές από 15 χώρε μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία και η Φιλανδία που έχουν υπευθυνθεί σχετική ερώτηση στην Επιτροπή. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η θέση σας. Ευχαριστώ. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντομπρόφσκης έχει το λόγο. Αγαπητά μέλη, θα ξεκινήσω με το θέμα της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας και των πίνακα αποτελεσμάτων και τι ακριβώς σημειώνουμε και τι χρειάζεται για να πάμε πιο γρήγορα. Οι αυξήσει στην έρευνα και στην ανάπτυξη εντάσσονται στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία παρακολουθούμε από πολύ κοντά στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Υπάρχουν χώρες οι οποίες συστηματικά εδώ μένουν πίσω και γι' αυτό εκδίδονται συστάσεις προς τις χώρες αυτές για την αύξηση της έρευνας των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη και επίση βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ε, δαπάνης σε συνεργασία με τις ε, βιομηχανικές δραστηριότητες. Για την ποιότητα τώρα των δημοσίων δαπανών. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σαφές στην ε, έκθεση ετήσιας ε, ανάπτυξης την οποία έχουμε εκδώσει και χαρακτηρίζει το σύνολο του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. για την απασχόληση και τις ανισότητες όπως αυτές ε, προσμετρούνται από τους δείκτες Τζένι. Είπα ότι το θέμα της ανισότητας είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε και αυτό μέσα από τη διαδικασία Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Προσπαθούμε να αυξήσουμε ε, τα επίπεδα ποιότητας των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας. Υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας όπως μέσω της φορολογικής πολιτικής όπως και έβρεση άλλων τρόπων μείωσης ε, των, της φορολογίας ε, της χαμηλά αμοιβόμενης απασχόλησης. Βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κοινωνικά συστήματα, βλέπουμε σε ποιο βαθμό είναι σωστά στοχευμένα στα τμήματα της κοινωνίας που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες, τις υψηλότερες ανάγκες Επίσης ασχολούμεθα και με το θέμα της κατάρτισης. Βλέπουμε πού υπάρχει υστέρηση στην σωστή κατάρχηση τμήματων του πληθυσμού που υπαρχει η στερηση στην σωστη αποκλεισμό από την απασχόληση. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βοηθήσουμε την ανισότητα που υπάρχει ε, στις αμοιβέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις επενδύσεις τώρα Πράγματι εμείς είδαμε ότι από το 2010 μέχρι το 2016 έχει υπάρξει πτώση στις επενδύσεις. Τώρα έχουν αρχίσει κάπως να αυξάνονται οι δημόσιες επενδύσεις. Περιμένουμε μία μικρή αύξηση για του χρόνου, αλλά είμαστε πολύ πιο χαμηλά από τα επίπεδα προκρίσεως και γι' αυτό ακριβώς εμένουμε τόσο πολύ στις επενδύσεις, είναι βασική μας προτεραιότητα. Σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Εμείς εκδώσαμε μία ανακοίνωση για την σωστή χρήση της ευελιξίας και μία από τις ρήτρες ε, του συμφώνου είναι η ρήτρα για τις επενδύσεις που δίνει την δυνατότητα στα κράτη-μέλη προσωρινά να αποκλίνουν από τον σεβασμό των ρυθμίσεων για να αυξήσουν τις επενδύσεις σε τομείς όπου αυτό είναι απαραίτητο. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει και εδώ δυνατότητα παρέμβασης στον τομέα τώρα της απασχόλησης μόνιμων θέσεων απασχόλησης, part-time επιμέρους απασχόλησης χρονικής, κυκλικής οικονομίας κτλ. Εδώ υπάρχουν τομείς στους οποίους θα πρέπει να γίνουν βήματα προόδου και στα πλαίσια των κανονισμών της Ένωσης, χωρίς να αγνοούμε τον βασικό μας στόχο, ο οποίος είναι κοινωνική προστασία για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να καλύπτονται κοινωνικά. Ο κύριος Μοσκοβισή να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Καλβέ Σομπό, μην ανησυχείτε, στα γαλλικά θα σας απαντήσω. Κατανοείτε πολλές γλώσσες κύριε Σομπό, αλλά λοιπόν ε, όλες οι ερωτήσεις που τέθηκαν στρέφονται στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Υπάρχουν τρία επίπεδα απάντησης σε αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω καταρχάς ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι οι επενδύσεις είναι χαμηλές λόγω του συμφώνου. Όχι, ίσα ίσα όλο και περισσότερο εμείς χρησιμοποιούμε το σύμφωνο όχι μόνο για να ελέγξουμε την δημόσια δαπάνη αλλά και να βελτιώσουμε την ποιότητά της. Εμείς ακριβώς κάνουμε τα λεγόμενα spending reviews σε διάφορες χώρες και έτσι προσπαθούμε να προετοιμάσουμε το μέλλον καλύτερα. Έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε και σε συγκεκριμένους τομείς, τομείς που είναι ιδιαίτεροι για σας, εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια, ε, πώς δηλαδή εμείς να συνδυάσουμε την ανθεκτικότητα με την ανάπτυξη. Λοιπόν, ποιοι είναι οι τρεις τομείς που θέλουμε να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις. Πρώτον, το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Εμείς ε, σε έφθετο χρόνο ε, θα καταθέσουμε τις συστάσεις μας άνα χώρα και θα δείτε ότι ε, θα στρέφουν την προσοχή μας στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Δεύτερον, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο προωθεί την έρευνα και την ανάπτυξη ήδη. Και τρίτον, είναι μια συζήτηση που θα γίνει πολύ σύντομα Πιστεύω πολύ στο μέλλον της σταθεροποιητικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής και Νομισματικής Ένωσης. Αυτό θα μας βοηθήσει να συντηρήσουμε ικανοποιητικά επίπεδα επενδύσεων σε περιπτώσεις εκ νέου ύφεσης ή οικονομικού ε, σοκ. Ε, τώρα η έλλειψη, αν θέλετε, το έλλειμμα το επενδυτικό είναι μια έννοια επί της οποίας εργάζεται η Ευρωπαϊκή εδώ και αρκετό χρόνο. Πράγματι δεν έχουμε ξαναφτάσει στα επίπεδα τα επενδυτικά πριν από την κρίση και επενδύουμε πολύ λιγότερο από τους ανταγωνιστές μας. Αν δεν είμαστε εδώ να έρθουμε ξανά στην κορυφή των επενδύσεων δεν θα παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία σε 5, 10 ή 15 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθεί και το πρόγραμμα Juncker των στρατηγικών επενδύσεων, μέσω κυρίως των ιδιωτικών επενδύσεων βέβαια, αλλά αναφέρεται και στο σύμφωνο σταθερότητας, το οποίο περιλαμβάνει μια ρήτρα επενδυτική, η οποία ήδη χρησιμοποιήθηκε για χώρες οι οποίες είναι στο προληπτικό επίπεδο Υπάρχει και η περίπτωση της Ισπανίας όπως είπατε που μπορεί να βγει από τη διαδικασία ελέγχου το επόμενο χρόνο, είναι σε οριακό επίπεδο στην φάση αυτή και νομίζω ότι το 18 αυτό θα είναι ξεκάθαρο σε σχέση με το υπερβολικό έλλειμμα και θα είναι επιλέξιμη για τη χρήση της ρήτρα αυτής και θα εξετάσουμε το αίτημα αυτό ανάλογα με τα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα έχουμε υπόψη. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Ε, θα περάσουμε τώρα στο τέταρτο γύρο να δώσουμε το λόγο στον Μπάς Άικελ από τους Πράσινους, ο οποίος εκπροσωπεί και την Έμπλ και την Econ. Έχει το λόγο για τρία λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεση αυτή, η οποία δίνει λίγο παραπάνω έμφαση στην φόρο διαφυγή, φόρο και στα ζητήματα κοινωνικής ε, δικαιοσύνης και ισότητας. Οπότε υπάρχει μια μικρή βελτίωση κατά τη γνώμη μας. Καλό είναι αυτό, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο στόχο μας. Ε, πολλά έχουν ήδη υποθεί για τι επενδύσει προ τον κύριο Χουτμάρκ να πω ότι συμφωνώ απολύτω. Ένα από τα προβλήματα είναι η έλλειψη επενδύσεων που τονίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω, όπω έχετε δει ότι αναφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα επίπεδα ε, ιδιωτικών επενδύσεων σε ονομαστικές αξίε είναι στα ε, επίπεδα πριν από την κρίση, Όμω το πρόβλημα είναι στι δημόσιε δαπάνε, τη συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όταν λέει η Επιτροπή λοιπόν πώ θα άρουμε τι θανοπού για τι επενδύσει. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς θα γίνει αυτό για τις δημόσιε δαπάνες, γιατί ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει ξανά και ξανά μόνο για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Έχετε κάνει κάποιες προτάσεις από αυτού, όμως για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ε, η έλλειψη δημοσιονομικού περιθωρίου για κάποιες ε, χώρε. Από την άλλη, εμένουμε στην ε, ουδέτερη δημοσιονομική στάση, το οποίο δημιουργεί ακριβώς ασφυξία. Ε, οπότε δεν ξέρω ακριβώς, αποφεύγει μάλλον η Επιτροπή να απαντήσει σε αυτό. Δεύτερον, φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή. Λέτε περισσότερο και αυτό είναι καλό. Όμω για τον κύριο Μοσκοβισή πιο συγκεκριμένα, ξέρουμε όλοι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι για την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ότι υπάρχει, ε, απαιτείται ομοφωνία στο Συμβούλιο. Ήδη έχετε πει στο Κοινοβούλιο στο παρελθόν ότι αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το άρθρο 116 της Συνθήκης Λισαβόνα, ε, πρέπει να καταλήξετε σε, να μας δώσετε μια ε, πρόταση ε, χρήσης ειδική πλειοψηφία για τα φορολογικά ζητήματα. Πότε θα έρθει αυτή η πρόταση και για ποιο ζήτημα, γιατί νομίζω ότι αυτή η συζήτηση στο να σπάσουμε τον κανόνα της ομόφωνης απόφασης για τα φορολογικά ζητήματα είναι κέρια σημασία για τη Θα ήθελα πιο συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτό. Μετά, για τα ζητήματα μακροοικονομικής ανισορροπίας. Αν δείτε τις βελτιώσεις που έχουν γίνει, έγιναν κατά κύριο λόγο στις χώρες που έχουν ελλείμματα. Οι χώρες με πλεονάσματα, ναι, συχνά αναφέρεστε στη Γερμανία, αλλά εκεί είναι κάτι χαμηλότερο από πέρσι. Αν το συγκρίνετε όμως μετά από πέντε χρόνια και πάλι έχει αυξηθεί το πλεόνασμά τους και στις κάτω χώρες. Δεν, έχουμε τα ίδια πλεονάσματα. Οπότε αν δείτε συνολικά την ανισορροπία, όλα είναι και περισσότερες χώρες στην Ευρώπη έχουν πλεόνασμα και το ερώτημα μου είναι πώς θα βελτιώσουμε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες για να έχουμε μεγαλύτερη ισορροπία στο μέλλον. Γιατί αυτή τη στιγμή ε, οι χώρες υπερχρεωμένες είναι αυτές που έχουν τελικά τα αποτελέσματα και όχι αυτές με τα πλεονάσματα. Γι' αυτό θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ευχαριστούμε κύριο, τον, τον κύριο Άικχαουτ ο κύριος Δομινίκη Μαχτά από το ΕΝΕΦ e στην Επιτροπή Απασχόλησης. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν είχατε μαζί ομιλία. Εγώ εκπλήσωμαι από την αυταρέσκεια που δείχνετε. και οι δύο όταν μα λέτε ότι έχει έρθει η ανάκαμψη, τα πράγματα πάνε καλύτερα μόνο και μόνο χάρη στι δικέ σα πολιτικέ. Εγώ θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι δεν είναι χάρη στι δικέ σα πολιτικέ. Πρόκειται για τη σύγκληση τριών ε, κριτηρίων που ε, σα εξυπηρετούν καθώ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πρόκειται για τα πολύ χαμηλά επιτόκια, πρόκειται για μια συνολική ανάκαμψη. Υπάρχουν λοιπόν άλλοι παράγοντε που δεν συνδέονται με δική σα πολιτική. Είναι το αποτέλεσμα των όσων συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη. Το ερώτημά μου... Νομίζω έχω 1,5 λεπτό διάθεσή μου, σωστά. Λοιπόν, όλα τα μέτρα σας, είτε πρόκειται για την κινητικότητα που αναφέρατε. Ουσιαστικά πρόκειται για θέμα τον ανταγωνισμό και εκρίζωση. Μιλάτε για σύγκληση και αναρμόνιση, πρόκειται ε, για αύξηση τη επισφάλεια. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει, λέτε, ουσιαστικά λιτότητα ε, σε όλε τι χώρε μα. Ε, και πιο συγκεκριμένα στρέφουμε λοιπόν προς τον κύριο Μοσκοβισή. Ξέρω ε, πόσο κοντά είστε στη Ρουμανία. Γνωρίζουμε ε, ότι οι πόροι που δίνονται στην Ρουμανία είναι κοντά 4 ε, δις ευρώ το χρόνο. Όμω, την περασμένη εβδομάδα ακούσαμε ότι για 4 εκατομμύρια ε, δολάρια αγόρασε η ρουμανική κυβέρνηση αμερικανικού πυράβλους. Θεωρείτε ότι αυτό είναι, μπορούμε να, το δεκτούμε ή ότι θα, θα επαναφέρετε τη Ρουμανία στην τάξη που παίρνει ευρωπαϊκά κονδύλια και με αυτά αγοράζει αμερικανικούς πυράβλους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντομπρόφσκης έχει το λόγο. Παρακαλώ. Λοιπόν, επανέρχομαι στο ζήτημα των δημοσίων επενδύσεων. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, βλέπουμε μία σταδιακή αύξηση και των ε, δημοσίων επενδύσεων Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε αυτή την τάση. Αυτό βέβαια άπτεται και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Υπάρχει και ρήτρα ε, σε σχέση με τις επενδύσεις που επιτρέπει στις ε, χώρες να αποκλίνουν από τους ε, στόχους για να αυξήσουν τα επίπεδα επενδύσεων. Και ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη αξιοποιούν αυτή τη ρήτρα. Και δεύτερον έχουμε την ε, σύνθεση των δημοσίων οικονομικών, όπου και πάλι ε, συνιστούμε ε, την τροποποίηση της σύνθεσης δημοσίων οικονομικών για να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις, στην έρευνα και κοινοτομία. Και όλα αυτά εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Βέβαια, πάντα με μια ισορροπημένη προσέγγιση πρέπει να τα εξετάζουμε αυτά τα πράγματα. Αφενό, πρέπει ε, να δώσουμε κίνητρα για την οικονομική ανάπτυξη, από την άλλη να διασφαλίσουμε την μακροχρόνια και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών μα. Και πράγματι, κάποια κράτη-μέλη έχουν πολύ ψηλά επίπεδα δημοσίου ε, χρέου που θα πρέπει να μειωθεί. Ε, για να προετοιμαστούμε και για Πιθανέ ε, μελλοντικέ οικονομικές αναταράξει που ελπίζουμε να μην υπάρξουν, αλλά ε, εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να αυξήσουμε την ε, αντοχή των οικονομιών μας. Μετά, για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής είναι κάτι το οποίο βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα μας και θα το θίξουμε και στη συνέχεια. Και σίγουρα και αυτό αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στις συστάσεις μας προς τα κράτη-μέλη για τρόπους αντιμετώπισης ε, της φοροδιαφυγής και βελτίωσης ε, της ε, συγκέντρωσης των φόρων, της ίσπραξης δηλαδή. Τώρα για τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών και τα πλεονάσματα σε Γερμανία και κάτω χώρες. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που φέτος και η Γερμανία και οι κάτω χώρες ε, θεωρείται ότι έχουν οικονομικές ε, ανισότητες και θα λάβουν αντίστοιχες συστάσεις για να μειώσουν τα πλεονάσματά τους. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που αυτές οι χώρες υπόκειται σε, σε βάθος ε, αναθεώρηση για να εξετάσουμε ακριβώς τις ανισότητες. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι ε, ακολουθούμε μια ισορροπημένη προσέγγιση, κοιτάζουμε και τα ελλείμματα και τα μεγάλα πλονάσματα όμως. Και στρεφόμαστε και σε αυτά τα κρατη Μετά, για την ευρύτερη, το ευρύτερο οικονομικό τοπίο και κατά πόσο μας ε, ικανοποιούν ε, οι σημερινές οικονομικές προβλέψεις. Πράγματι είναι θετικές και εδώ και παγκοσμίω. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει μόνο να λέμε ότι μας ικανοποιεί η σημερινή κατάσταση, αλλά να αυξήσουμε, να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των οικονομιών μα και να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για ε, πιθανούς οικονομικούς κραδασμούς. Αυτό τονίζουμε και στην ε, ετήσια έκθεση προόδου, ότι πρέπει να παραμείνουμε στην τροχιά που έχουμε ε, χαράξει και ότι δεν μπορούμε να φυσικάζουμε. Ευχαριστούμε. Ο λόγο στην κυρία Μουσκοβισή. Ορισμένες ε, παρατηρήσεις από πλευρά μου. Πρώτον, ε, για την φορολογία. Πράγματι, δεν ε, μπορούμε ε, να εξετάζουμε και τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής και των δημοσιονομικών ζητημάτων εφόσον υπάρχει η απέτηση της ομοφωνίας. Είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να δημιουργεί προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε να το ε, αποφύγουμε και ε, ξέρω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού, γιατί αυτό ζητούν και οι πολίτες μας. Όμως πιστεύω ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ πολύ σωστά είπε στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ότι πρέπει να αλλάξει ακριβώς αυτός ο κανόνας. Δεν αγνοώ και αυτή την ρήτρα της ε, μεταβατικής ε, κατάστασης. Για να σας δώσω συγκεκριμένη απάντηση, εμείς ε, δεν έχουμε το μαγικό ραβδάκι. Πρόκειται για μια συλλογική πίεση που θα επιτρέψει μια σημαντική αλλαγή των πραγμάτων. Όμως, Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και απολύτως αδύναμοι απέναντι στην φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Ε, ήδη έχουμε κάνει πολλά. Πρέπει να το γνωρίσουμε αυτό. Και αυτό το σίγουρα το ξέρουν και τα μέλη της Επιτροπής ε, για τα έγγραφα του Παναμά. Έχουμε κάνει περισσότερα τώρα από την τελευταία τρία κονταετία. Ε, έχουμε πολλές διαφορετικές ε, νομοθετικές ρυθμίσεις, ε, country by country reporting που είναι δημόσιες και διαφανείς. Ε, για την πρόταση ενοποίησης της φορολογικής βάσης των επιχειρήσεων και πάλι βέβαια έχουμε περιθώριο βελτίωσης και ανάληψης δράσης και μπορούμε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματά μας με θεματικό τρόπο. Σε ό,τι φορά τις μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες, διαπιστώνουμε ότι ε, λίγες είναι οι μειώσεις που αναμένονται στη Γερμανία, στις κατοχώρες και στη Δανία. Υπάρχει λοιπόν μια συμμετρία, πρέπει να βρούμε μια ε, λύση και η σύσταση για την Ευρωζώνη, αλλά και οι συστάσεις μας, οι διοικές αναχώρας συστάσεις, προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Και πάλι όμως τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε ό,τι αφορά εμείς ε, συνεχώς ε, τα υπογραμμίζουμε και αναφέρουμε ότι υπάρχουν ε, συμμετρικές ανισότητες και ανισορροπίες μάλλον. Σε ό,τι αφορά τον εκπρόσωπο της άκρας δεξιάς, να αναφέρω... Εντάξει, θα προσπαθήσω να είμαι μετριοπαθής, ακόμα και αν κάθε φορά ταράζομαι. Δά, δεν είστε άκρα δεξιά, όλοι γνωρίζουν πως είστε. Σχόλια εκτός μικροφώνου. όχι στις προσωπικά πιστεύω, λέει ο Επίτροπο. όμω επί τη ουσίας να σταθώ. Είπατε ότι η ανάκαμψη δεν οφείλεται καθόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μόνο σε εξωτερικούς παράγοντες. Όλα αυτά είναι ανοησίες και σφάλματα. Ε, δεν λέω βέβαια ότι η ανάκαμψη οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στι ενέργειε Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι παράλογο να λέει κανεί ότι ε, δεν υπήρχε κανένα όφελο από τι ε, ευρωπαϊκέ ενέργειε. Γιατί πρόκειται για πράξει και προσπάθειε των ίδιων των Ευρωπαίων για να μειώσουν τα ελλείμματα, να ε, αναδιαρθρώσουν τι οικονομίε, να τι κάνουν πιο ελκυστικέ. Το οποίο θα μας, θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα και με την ανάκαμψη και εσείς ε, εμένετε σε μια προσέγγιση που αρνείται ακόμα και αυτά που λειτουργούν ε, καλά. Και αυτό δεν ε, ωφελεί ούτε τους Ευρωπαίους πολίτες ούτε κανέναν. υπάρχει και εδώ μία μικρή νότα μυσαλλοδοξίας που αναφέρατε ότι είμαι κοντά στη Ρουμανία. Ο πατέρας μου γεννήθηκε λοιπόν εκεί και είχε διωχθεί λόγω της θρησκείας του, αναγκάστηκε να διαφύγει. αυτό βέβαια ε, δεν σημαίνει ότι εγώ ήμουν ε, μεροληπτούσα όταν ζητούσα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι που μπήκε. Η Ρουμανία δεν είναι προτεκτοράτο, αγαπητέ κύριε. Είναι ε, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα. Και δεν είναι μοναδική χώρα που κάνει τέτοιες αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ε, πρέπει, αν δείτε τη γνώμη μας ε, σε αυτά τα ζητήματα, θα δείτε ότι εξετάζουμε σε ζητήματα ε, όπως είναι η αύξηση των ελλημάτων στη Ρουμανία και ζητούμε από την κυβέρνηση να τα ελέγξει. Αυτά μπορώ να σας πω σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη μας παρουσιάσατε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Επιτροπέ. Και τώρα να ακούσουμε την κυρία Σάνδρου. Εξ ονόματος του ΕΛΚ από την Επιτροπή Απασχόλησης. Πέμπτος γύρος ε, ερωταπαντήσεων. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Και εγώ θα ήθελα να πω, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ότι είμαι ικανοποιημένη που βλέπω που οι δείκτες, ότι οι δείκτες, ε, οι οικονομικοί δείκτες ε, παίρνουν τα πάνω τους ιδιαίτερος χάρη ε, στις προσπάθειες των Ευρωπαίων. Βλέπουμε λοιπόν ότι μειώνονται τα ελλείμματα, έχουμε οικονομική ανάπτυξη και ότι η ανεργία μειώνεται στο σύνολό τη. Ωστόσο, είναι θετικές αυτές οι εξέλιξεις ασφαλώς, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και διαφοροποιήσεις και ότι οι διαφορές είναι σημαντικές από κράτος μέλος, σε κράτος μέλος, από περιφέρεια σε περιφέρεια και μεταξύ κάποιων κατηγοριών του κόσμου διάφορες, ε, στις διάφορες ηλικίε, ε, στα διάφορα επαγγέλματα. Θα πρέπει λοιπόν να πιστεύω να καταβάλουμε ακόμα και άλλες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα πάει χέρι, χέρι, με χέρι με μια, οικονομική, με μια κοινωνική πραγματικά ανάκαμψη. Πώς θα φροντίσουμε λοιπόν να υπάρξει καλύτερος συντονισμός μεταξύ της οικονομικής πολιτικής και της κοινωνικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα. Υπάρχει κάποια εγκύτητα μεταξύ των ε, συμβουλίων της, ε, του ΕΚΟΦΗΝ και των ε, αντίστοιχων πολιτικών για τα κοινωνικά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα ζητήματα αυτά που έχουν μεγάλες επιπτώσεις και στους πολιτές και στις επιχειρήσεις. Αναρωτιέμαι μεταξύ των συγκεκριμένων συστάσεων αναχώρα για το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προβλέψει ιδιαίτερη θέση για τις εργατικές μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας στα κράτη-μέλη, σε ό,τι αφορά και την ψηφιακή εποχή που ζούμε. Ευχαριστούμε η κυρία Κάπελ από το ΙΕΝΑΦ, από την Επιτροπή Οίκων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους Επιτρόπους για τις εκθέσεις, για τις οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν και διάφοροι θετικοί δείκτες σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, τη μείωση της ενεργείας, αλλά φυσικά και μία αύξηση των επενδύσεων. Γιατί, όπως ακούσαμε, όμως παρόλα αυτά οι επενδύσεις δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο πριν από την κρίση. Και φυσικά δεν υπάρχει ακόμα ασφαλώς σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών. Είμαστε, απέχουμε παρασάγκα από την σύγκληση αυτή την επιθυμητή. Δύο είναι οι συστάσεις της Επιτροπής. Τα κράτη-μέλη με τα υψηλότερη χρέωση να προσέξουν σε ό,τι αφορά την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και τα κράτη-μέλη με πλεόνασμα σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητά τους θα πρέπει να προβούν σε επενδύσεις για να τονώσουν την ε, εσωτερική ζήτηση. Και θα πρέπει το δυναμικό παραγωγικότητας και ανάπτυξης να εξατληθεί, είπε ο Επίτροπος Ντρομπρόσκης. Ε, να επισημάνω στο, στο σημείο αυτό ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων για να μην δημιουργηθούν φούσκες. Προβλέπετε λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα για την καλύτερη κατανομή των πόρων και τον έλεγχο αυτής. Για παράδειγμα, στην ετήσια έκθεση για την αγωνιστικότητα του 2016 μιλάμε για τα ghost airports, ε, για αεροδρόμια, φαντάσματα. Έχετε εδώ πέρα μέσα για να πετύχετε την καλύτερη κατανομή των πόρων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ εκπροσωπεί το ΕΛΚ στην Επιτροπή ΕΛΚ Εικόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Έχω για σας, ε, κύριε Μοσκοβίση, μία ερώτηση σε ό,τι αφορά την ιδιωτική αγορά χρεών. Προφανώς η υπερχρέωση του κλάδου επισημαίνεται και στην μηχανισμό επαγρύπνησης και αυτή η υπερχρέωση ανάλογα και από τα κράτη-μέλη οφείλεται στην ε, μεγαλύτερη ε, χορηγήση ε, δανείων, Κυρίω ενυπόθηκων. Και στην Βέλγια έχουμε το θέμα αυτό. Και το κίνδυνο δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τα ακίνητα και την αξιολόγηση τους, αλλά με το πώ χρηματοδοτούν οι οικογένειε στην αγορά ενό ακινήτου. Και η Εθνική Μα Τράπεζα δημοσίευσε μια έκθεση που φαίνεται ότι θα ζητούσαμε έξτρα buffer κεφαλαίων για την ε, διατήρηση της ε, ανυπόθηκης αγοράς μας και πώς θα προσπαθήσουμε λοιπόν να λάβουμε υπόψη και να συνυπολογίσουμε αυτή την υπερχρέωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριοι Επίτροποι, θα δεχτείτε ε, από δύο μέλη ερωτήσεις ε, ενός λεπτού. Θα είστε προφανώς πολύ σύντομοι και στις απαντήσεις σας. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μαρία Ρένα, λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Μία ερώτηση σε ό,τι αφορά του ποσοστού, το ποσοστό ε, απασχόλησης και την ενεργεία και βλέπουμε ε, ότι δεν ε, ότι μιλάμε για αύξηση του όγκου α, της απασχόλησης. Τι ποιότητα όμως είναι οι θέσεις αυτές. Και μία δεύτερη ερώτηση για την απασχόληση. Το είδος, ε, για παράδειγμα, ε, οι γυναίκες θεωρούμε ότι ε, συμμετέχουν στην αύξηση της αποσχολησιμότητας ε, σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Το δείξατε αυτό και το βλέπω και στην έκθεσή σας ότι θα δώσει πιο πολύ προσοχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κόστος εργασίας σε κάποιες χώρες όπως η Ουγγαρία, η Λουθουανία και το καθεξής η Λετωνία. Τι, θα, τι σημαίνει όμως αυτό, ότι θα ζητήσετε από τις χώρες αυτές να μειώσουν το μισθολογικό κόστος ενώ ουσιαστικά θέλουμε σύγκληση και υπάρχουν μεγάλες διαφορές μισθολογικές μεταξύ των χωρών αυτών και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάει προς τη σωστή κατεύθυνση λοιπόν η εξέλιξη του μισθολογικού κόστους. Και ο κύριος Πάβελ, τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και επιτροπή που είσαστε εδώ σήμερα. Πολλά θέματα θέλω να δείξω, εν πάση περιπτώσει θα περιοριστώ για την χώρα μου, τη Ρουμανία. Στις αρχές του έτους φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την εκτίμηση ότι ήμασταν πολύ πιο κάτω από ό,τι προκύπτει στην πράξη ότι βρισκόμαστε στα τέλη του ε, έτους. 5,6 έχουμε λοιπόν τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 6,1% και 6,5% εκτιμά το Moody's ε, την κατάστασή μας. Λέτε λοιπόν στην έκθεση ότι το μακροπρόθεσμα η ανάπτυξη αυτή δεν είναι βιώσιμη και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το έλλειμμα. Αλλά η εκτίμηση της κυβέρνησης είναι ότι το έλλειμμα θα μείνει στο 2,6%. Το χειρότερο θεωρώ. Μάλλον, δεν χρησιμοποιούνται καλά επιχειρήματα. Η αύξηση αυτή δεν οφείλεται μόνο στην ιστορική κατανόληση, αλλά επειδή η βιομηχανία μας αυξάνεται 7,7% και η εσωτερική κατανάλωση και η γεωργία και το ICT. Πείτε μας λοιπόν τι σας απασχολεί πραγματικά στην περίπτωσή μας και πώς μπορούμε να έχουμε εκτιμήσεις και αξιολογήσεις πιο κοντά στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τη Ρουμανία γιατί δεν κάνει καλό. Πραγματικά δεν μας ωφελεί αυτή η μεγάλη διαφορά. Ευχαριστώ παρολί. Τέσσερις ερωτήσεις ε, και να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, για το πώς ε, μπορούμε να βελτιώσουμε τις οικονομικές και πολιτικές ε, και κοινωνικές πολιτικές μας. Από την έναρξη της θητείας μας είχαμε ξεκαθαρίσει ότι εξετάζαμε τις οικονομικές και δημοσιονομικές, κοινωνικές και εργασιακέ προκλήσεις. Όλα αυτά λοιπόν τα συνεξετάζαμε. Θεωρούσαμε ότι είναι αλληλένδετα και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και πάλι τα συνυπολογίζουμε για να σας ε, δώσω μια εικόνα. Το 40% των ε, ειδικών αναχώραση στάσεων που απευθύνουμε στα κράτη-μέλη συνδέονται με κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα. Και αυτή η τάση θα ενισχυθεί στο μέλλον καθώς θα λαμβάνουμε υπόψη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σε ό,τι αφορά τώρα την ψηφιακή οικονομία, έχουμε και την πρωτοβουλία μας για την ενιαία ψηφιακή αγορά, έχουμε και ένα ψηφιακό, μάλλον θεματολόγιο ψηφιακών δεξιοτήτων είναι σαφές ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις δεξιότητες της αγοράς εργασίας στην ψηφιακή οικονομία. Και υπάρχει σημαντικό έλλειμμα και χάσμα ε, ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά και το θέμα των επενδύσεων και τη σύγκληση των ε, μισθών, αποτελεσματική χρήση των πόρων. Σε το φορά τη σύγκληση λοιπόν, πράγματι, μεταξύ των κρατών μελών. Για παράδειγμα, στην Ευρωζώνη βλέπουμε ότι η σύγκληση αυτή καθυστερεί μετά την κρίση. Έχει σταματήσει και τώρα προσπαθούμε να επανεκκινήσουμε αυτή τη διαδικασία της σύγκλησης. Αυτό αποτελεί τμήμα του θεματολογίου μας στο ψηφιακό εξάμεινο ε, και θα εμπεριέχεται και στις προτάσεις μας για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σε ό,τι αφορά τώρα την αποτελεσματική χρήση και κατανομή των πόρων είναι κάτι το έχουμε λάβει υπόψη ε, σε ό,τι αφορά τη σύνθεση και την ποιότητα των δημοσίων οικονομικών. Τώρα, εξελίξεις στην αγορά κινήτων και για τα ανυπόθηκα δάνεια και αυτά τα παρακολουθούμε και το Ευρωπαϊκό ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συστημικών Κινδύνων έχει εκδώσει ειδοποιήσει σε ό,τι αφορά την, εξελίξει εξελίξεις αγορέ ακινήτων και παρακολουθούμε τις εξελίξεις ε, και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου υπάρχουν ειδικέ συστάσεις λοιπόν για να αποφύγουμε την ε, τη δημιουργία φούσκας σε συγκεκριμένες ε, αγορές. Τώρα, για το ποσοστό της απασχόλησης μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε ιστορικά υψηλά ε, σε ό,τι αφορά την απασχόληση. και με συνεχώς αυξητικές τάσεις. Βέβαια, έχουμε περισσότερη μερική απασχόληση και διάφορες νέες μορφές απασχόλησης. Γι' αυτό και τονίζουμε ότι και σε αυτές τις θέσεις εργασίας θα πρέπει να διασφαλίζεται η κοινωνική προστασία των εργαζομένων. Και αυτός είναι και ο σκοπός της πρωτοβουλίας μας, η ε, κοινωνική προστασία για όλους. Τώρα, για το ε, χάσμα μεταξύ των φύλων, στην απασχόληση και στους μισθούς, αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν ε, ε, κάποιες χώρες οποίε το πρόβλημα αυτό είναι πιο έντονο ακόμα. Για τη Ρουμανία... Πράγματι αναμένεται ανάπτυξη της τάξης του 5,7% είναι από τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, όμως έχουμε και, το, και μεγάλη αύξηση του ελλείμματος. Το 2015 ήταν 18%, πέρσι ήταν 3%, φέτος περιμένουμε πάλι 3% περίπου και του χρόνου, αν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, 3,9% ήδη το έλλειμμα επί του ΑΕΠ. Υπάρχει λοιπόν σημαντική απόκληση από τον ε, ε, μεσοπρόθεσμο στόχο, γι' αυτό και η Ρουμανία για τη Ρουμανία έχουμε κινητοποιήσει τις σχετικές ε, διαδικασίες υπό το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Μοσκοβισή τώρα έχει το λόγο. Ο συνάδελφος ε, απάντησε στα περισσότερα. Θα ήθελα μόνο να επιμείνω στην γεγονό ότι σε κάποια κράτη-μέλη Υπάρχουν κάποιες ανησυχητικέ ενδείξεις, ιδίως ό,τι αφορά τις αγορές ακινήτων στη Σουηδία, στην Αυστρία, Δανία, Λουξεμβούργο, κάτω χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί υπάρχουν σημαντικές πιέσεις ε, στις τιμές, ιδίως στον ε, τομέα των ακινήτων και με υψηλά επίπεδα ε, ιδιωτικού δανεισμού και εδώ θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν διορθώσεις σε αυτές τις χώρες τουλάχιστον. Για τη Ρουμανία. Έχω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, για την ανάπτυξη που πράγματι υπάρχει στην ε, Ρουμανία, σημαντική ανάπτυξη. Τώρα πρέπει να δούμε αν θα είναι διαρκής και μακροχρόνια. Πρέπει να το δούμε αυτό με μεγάλη προσοχή. Θετικό βέβαια είναι που πηγαίνει καλά οικονομικά αυτή η χώρα, όμως και πάλι πρέπει να εξετάζουμε τους ε, παράγοντες ανάπτυξης για να σιγουρευτούμε ότι θα είναι όντως μόνιμη αυτή και βιώσιμη αυτή η ανάπτυξη. Το πιο σημαντικό όμως εδώ που αναφέρθηκε ήταν τα δημόσια οικονομικά. Με τόσο σημαντική ανάπτυξη, το λογικό είναι το έλλειμμα της Ρουμανίας να συρρυκνωθεί και μάλιστα γρήγορα. Ενώ εμείς βλέπουμε το αντίθετο. Σκοπός αυτής της ε, διαδικασίας σημαντικής απόκλησης είναι να ενθαρρύνουμε αυτό το κράτος μέλος να επιστρέψει στον δρόμο ε, της ε, βελτίωσης και για να αποφύγουμε τη διολίστηση προς ένα υπερβολικό έλλειμμα. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του 1466 του 97 κανονισμού, η Επιτροπή απευθύνει τέτοιες συστάσεις για την αντιμετώπιση ε, της ε, σημαντικής αυτής απόκλησης. Επικεντρωνόμαστε στο 2018, δεδομένη της επιπλέον ε, διολύσεις του 2017. Η απόσταση είναι ακόμα μεγαλύτερη σχέση με την άνοιξη του 2017, οπότε πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να επιστρέψουμε στην σόφρονα δημοσιονομική πολιτική και αυτό μάλιστα κατεπηγόντως εάν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι ναι, είναι τόσο σημαντική η οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και ε, ασκούμε πιέσεις προς τη Ρουμανία να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για ε, να επιστρέψει στις συνήθεις διαδικασίες και έτσι να ξεφύγει από την διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος. Okay, thank you. Um, I think we stop there. Uh, Εντάξει, θα μείνουμε εδώ. Τι είναι εδώ αυτός ο γύρος ερωταπαντήσεων. Μπορούμε να πούμε μόνο ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα και όλοι το ξέρουμε αυτό όμως έχουμε επιστρέψει στον ίσιο δρόμο. Και αυτό είναι μια καλή αφετηρία. Όταν απευθυνθούμε και στους ε, ψηφοφόρους μας του χρόνου. Ευχαριστούμε τους ε, δύο επιτρόπους. Ευχαριστούμε και τις δύο επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Απασχόλησης. και σίγουρα θα υπάρξουν τέτοιες συζητήσεις και στο μέλλον στις δύο επιτροπές μας για να βρούμε συγκεκριμένε λύσεις για το μέλλον. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας.